Ε, άποψη της Επιτροπής η οποία με αποτέλεσμα 21 προς 13 τάχθηκε υπέρ του ψηφίσματός μας. Ακούστε, ήταν ε, συμφωνία. Ε, ο κύριος Μπράιαν Σίμψον συμφώνησε. One uh, Έχω μια πρόταση ψηφίσματος στο τέλος της συζήτησης από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, χωρίς μικρόφωνο ο κύριος Κράμερ. Και πάλι ε, με ενημέρωσαν ότι υπήρξε συμφωνία στην Επιτροπή. Συζητήστε το άλλη φορά ή συζητήστε το στην Επιτροπή. Δεν είναι δική μου δουλειά. Ε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έκλεισε η συζήτηση. Αύριο στις 11.30 θα ψηφίσουμε. Το επόμενο σημείο είναι μια προφορική ερώτηση εφαρμογή του κανονισμού REMIT και προπολογισμό του οργανισμού ASER για το 2014. Πρώτη ομιλήτρια η κυρία ε, Ρωμάνα Τζόρνταν που είναι η συγκήτρια αυτή της, ε, αυτής της ερώτησης. Πριν από το τέλος ε, το μέσο, μέσα της επόμενης ε, χρονιά θα πρέπει να δημιουργήσουμε την εσωτερική αγορά και έχουμε ε, προχωρήσει με την αποστολή μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κανονισμός REMIT προβλέπει ότι ο ACER, ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, πρέπει να αναλύσει την αγορά ε, ηλεκτρισμού και αερίου και οποιασδήποτε παρεμβιάσεις της ε, νομοθεσίας και καταχρήσεις. Ο κανονισμός αυτός, ε, με τον κανονισμό αυτό θα πρέπει να διασφαλίσουμε μια στενή συνεργασία. Για να το κάνουμε αυτό, ο Acer χρειάζεται πόρους, χρηματικούς πόρους και ε, ανθρώπινους πόρους και θα πρέπει να δημιουργήσει, ε, να υπάρξει υψηλή εμπιστοσύνη στον Acer. Το 2012 ο οργανισμός είχε επαρκή πόρους. Ο προπολογισμός ε, ο φετινός είναι χαμηλότερος κατά 3 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόβλημα επιδεινώνεται συνεχώς διότι η Επιτροπή για το 2014 προβλέπει περίπου 5 ε, εκατομμύρια ευρώ λιγότερα στον προπολογισμό από αυτά που χρειάζεται ο οργανισμός. Το πρόβλημα είναι ακόμη πιο οξύ γιατί στην ουσία δεν θα καλυφθούν επιπρόσθετες θέσεις απασχόλησης, ενώ χρειάζονται περίπου 50 πρόσθετοι υπάλληλοι. Ε, ο Acer δεν θα μπορέσει να αγοράσει τον εξοπλισμό που χρειάζεται, τον απαιτούμενο ε, εξοπλισμό που χρειάζεται και αυτό είναι ανησυχητικό. Σύμφωνα με τις ε, πληροφορίες που έχουμε λάβει, το ε, σχέδιο προπολογισμού δεν προβλέπει ούτε την εκτέλεση των αποστολών του οργανισμού που είναι απαραίτητες. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες από αυτές τις αποστολές είναι δημιουργία ε, ενός μητρού ε, των ε, συμμετεχόνων στην αγορά ενέργειας, την θέσπιση στενών σχέσεων ανάμεσα σε οργανώσεις αγοράς, τη δημοσίευση των δεδομένων του Acer και επίσης δεδομένα που αφορούν αυτούς που ασχολούνται σε επιστημονικό επίπεδο και πιο στενή συνεργασία με άλλους φορείς όπως η ΕΣΜΑ. Οι εκπρόσωποι του οργανισμού εξέφρασαν τις ανησυχίες του. Εάν ο δεν θα μπορέσει να εκπληρώσει τα καθήκοντά του και την αποστολή του θα είναι ο νόμος της ζούγκλας. Κανείς δεν θα μπορέσει να συγκεντρώσει τα στοιχεία, να τα αναλύσει ε, για να προλάβει τις καταχρήσεις και την απάτη. Και γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι η μη υλοποίηση των διατάξεων του κανονισμού REMIT θα μπορούσε να δικαιοδεύσει τη διαφάνεια και την ακεραιότητα της αγοράς μας, της αγοράς ενέργειας, ε, ηλεκτρισμού και ε, αερίου και ως αποτέλεσμα αυτό ε, θα έχει επίπτωση και στις τιμές ενέργειας. Θα ήθελα επίσης να θέσω τα ακόλουθα ερωτήματα πώς ε, θέλουμε να πετύχουμε την εσωτερική αγορά της ενέργειας, ηλεκτρισμού και αερίου. Ε, με την ε, αλλαγή του προπολογισμού για το 2003 θα μπορέσουμε να έχουμε την αγορά απαιτούμενου εξοπλισμού και πώς ο ΕΙΣΕ θα μπορέσει να αγοράσει αυτό τον εξοπλισμό χωρίς να αλλάξει ο προπολογισμός του 2013. Και η Κομισιόν είναι διατεθειμένη να εγκρίνει ένα σοβαρό προπολογισμό για το 2014 που να μην διακυβεύει την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Κυρίες και κύριοι, αυτά θα μπορούσαν να δημιουργήσουν περισσότερες ζημιές και εντός της ε, Επιτροπής ΙΤΡΕ είμαστε πεπισμένοι ότι χρειάζεται ένα επίπεδο ε, ε, επαρκούς χρηματοδότησης για τον οργανισμό Acer, για το καλό των Ευρωπαίων καταναλωτών. Να καλωσορίσω τον Επίτροπο Έντιγκερ και να του δώσω το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, Ε, είμαι ευγνώμων στη συνάδελφο που παρακολούθησε τη λειτουργία του οργανισμού και θέτει και θεμητά ερωτήματα για τη λειτουργία του. Ο Άσερ είναι νεαρός οργανισμός. Εδώ και δύο χρόνια έχει κι άλλο ένα καθήκον, δηλαδή να ελέγχει την ε, ε, μεγάλη αγορά ενέργειας και να παρεμποδίζει καταχρηστικές ε, πρακτικές και να τις απαγορεύει. Πρέπει να παρακολουθεί την αγορά, να ε, εκδίδει ε, προδιαγραφές σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας. Ο ΆΣΕΡ έχει γι' αυτό εξοπλισμό επεξεργασίας δεδομένων που πρέπει να ανταποκρίνονται σε πρότυπα προστασίας δεδομένων. Στα πλαίσια του προϋπολογισμού του 2013 διαθέσαμε από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ποσά για τον ΑΣΕΡ, για την αγορά λογισμικού και υπολογιστών. Ε, αυτές οι ανάγκες καλύφθηκαν. Ε, θα πρέπει όμως και η αρχή του προϋπολογισμού να εγκρίνει τις δαπάνες που προβλέπονται για αυτό το έτος. Διαβεβαιώνω ότι και για το 2014 στα πλαίσια της απόφασης για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα υπάρχει πρόνοια για τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων και, για όλη την... και έχουμε προβλέψει κονδύλια για το κομμάτι της τεχνολογίας της πληροφορίας. Ε, αγορά λογισμικού, υπολογιστών και θέση σε λειτουργία όλων αυτών. Ε, χρειαζόμαστε όμως και εργαζομένους. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει και το κατάλληλο ειδικευμένο προσωπικό. Γι' αυτό έχουμε δημιουργήσει 15 θέσεις εργασίας που έχουν καλυφθεί από τον οργανισμό. Πιστεύουμε ότι το 2014 θα επαρκούν τα διαθέσιμα κονδύλια για την κάλυψη αυτών των δαπανών αν χρειαστούν ε, ε, περισσότερα θα, τα, θα επεξεργαστούμε τα σχετικά αιτήματα και ανάγκες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά η Κομισιόν και οι υπηρεσίες της ε, θα πρέπει να μειώνουν κάθε χρόνο κατά 1% σε 5 χρόνια 5% το προσωπικό και αυτό ε, ισχύει όπως και για τα κράτη-μέλη. Θα... Με τον Άσερ αρχίσαμε και μία άλλη διαδικασία, δηλαδή τα δημοσιονομικά κονδύλια να δοθούν κατά προτεραιότητα στην εφαρμογή του κανονισμού REMIT ε, μέσα στον Άσερ γίνονται κάποιες αναδιαρθρώσεις δηλαδή και τις παρακολουθούμε. Σας διαβεβαιώνω ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ο κανονισμός REMIT προτάθηκε από μας ε, με σκοπό να επιτύχει και τον παρακολουθούμε ούτως ώστε να υπάρχει διαφάνεια στην αγορά εργασίας και πλεονεκτήματα για τους πολίτες ε, δηλαδή να μην γίνονται καταχρήσεις και να είναι και ικανοποιητικές οι τιμές ενέργειας. Ε, σας ε, ευχαριστώ πολύ και είμαι διατεθειμένος να βοηθήσω για την περαιτέρω υλοποίηση του κανονισμού. Καλά. Ευχαριστώ πολύ, ε, κυρία Μάτσε Κούκοβιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε Έτιγκερ. Αν ε, είμαστε σοβαροί όταν μιλάμε για την εσωτερική αγορά, Βεβαίως ε, η αγορά ενέργειας είναι ένα από τους πυλώνες αυτής της αγοράς και ο Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Ερχών Ενέργειας, ο ΆΣΕΡ, ε, έχει την έδρα του στη Σλοβενία και ένας από τους λίγους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και μπορώ να σας πω ότι ε, δυστυχώς αυτά που συμβαίνουν έχουν, έχουν οδηγήσει σε αύξηση του ευρωσκεπτικισμού. Πώς μπορούν να υπάρχουν ε, τόσο μεγάλες διαφορές σε σχέση ε, με τις ανάγκες, δηλαδή τόσο αποκλίνουσες απόψεις σε σχέση με το απαραίτητο προσωπικό και την απαραίτητη χρηματοδότηση. Και αναρωτιέμαι, αν είμαστε πράγματι σοβαροί και τι θέλουμε να κάνουμε με αυτόν τον οργανισμό. Αν πράγματι εμείς στην Ευρώπη θέλουμε να εποπτεύουμε την αγορά ενέργειας και αν θέλουμε να έχουμε χαμηλότερο κόστος αν ε, δούμε το ποσό που προβλέπεται ως ε, επένδυση, τα 200 εκατομμύρια ευρώ που προβλέπονται για την υποδομή, τα κονδύλια για τον Άσερ είναι πραγματικά ένα πολύ μικρό μέρος αυτού του ποσού και δεδομένης της κρίσης ε, είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μειώσουμε και τον ευρωσκεπτικισμό. Ευχαριστώ κύριε Σκορίεντε Κάπος για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, που παρευρίσκεστε στη συζήτηση αυτή η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας εξαρτάται από υποδομές και από σύγχρονες διασυνδέσεις περιβαλλοντικής εφορίας κοινών προτύπων, ενερμονισμένων κανόνων και πρέπει να είναι ε, ανταγωνιστικός και διαφανής σε όλους αυτούς ε, τους τομείς, ε, σε ο Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Έρχων Ενέργειας διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην εφαρμογή του κανονισμού για τις υποδομές, την παρακολούθηση των αγορών ενέργειας, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια, κανονισμός REMIT, στην εφαρμογή του τρίτου ενεργειακού πακέτου και στον καθορισμό των κωδικών δικτύων, ε, η εφαρμογή των πολιτικών θέλει ε, να μπορεί να υλοποιεί ο Άσερ τα καθήκοντά του. Όμως ε, η Κομισιόν προτείνει περικοπή ένα τρίτο περίπου φτάνουμε στα 11 εκατομμύρια ευρώ και είναι πραγματικά εκπληκτική η απόσταση που υπάρχει μεταξύ ε, των φιλοδοξιών ε, θεωρητικά ε, για να έχουμε μια ενεργειακή αγορά και των μειοπικών αποφάσεων. Δεν είναι μόνο το 2014 που διακυβεύεται εδώ. Μετά από το 2014 θα έχουμε μια νέα κομισιόν, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και το μέλλον με μη κατάλληλα μέσα και λυπής λύσεις και αν υπερισχύουν οι εθνικές λογικές για την ενεργειακή πολιτική, θα οδηγηθούμε σε απελπισία. Δηλαδή γλιτώνουμε 5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ε, ε, ε τίθενται πάρα πολύ κίνδυνοι και θα οδηγηθούμε σε απώλεια παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας ε, και θα έχουμε με τα εγκατάσταση των επιχειρήσεων και περισσότερων περισσότερη ενεργεία στην Ευρώπη. Δεν είναι αυτό όμω που θέλει η Κομισιόν, φαντάζομαι. Η Ευρώπη χρειάζεται πολύ καλύτερε αποφάσει. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ε, υπάρχει ενδιαφέρον ε, για το Catch the Eye. Και έτσι λοιπόν θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο Έντιγκερ για κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις. Ich kann Ihren Argumenten, dass wir eine starke Behörde brauchen, dass wir Βεβαίως χρειαζόμαστε έναν ισχυρό οργανισμό για την εφαρμογή του REMIT, θα πρέπει η αγορά να ολοκληρωθεί, ε, θα πρέπει να επιτηρούμε ε, ώστε να εφαρμόζονται σωστά καμία αντίρρηση εδώ ε, και μπορεί να χρειαστούν και άλλες θέσεις εργασίας. Ε, όμως στα πλαίσια των ε, διαβουλεύσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και για το, πολυε, το ε, δημοσιονομικό πλαίσιο έχουμε, ε, ένα στενό, έχουμε αποφασίσει για ένα στενό προϋπολογισμό. έχουμε, όπως σας είπα, πρόγραμμα μείωσης 5% σε 5 χρόνια. Ε, ενδεχομένως θα θέλαμε κάτι διαφορετικό ε, εάν υπάρχουν εδώ ε, εξαιρέσεις, αυτό σημαίνει ότι άλλοι οργανισμοί ή αντιπροσωπείες ε, σε άλλες χώρες θα πρέπει να μειωθούν πολύ περισσότερο. Και αυτό δεν θα βρει σύμφωνους τους συναδέλφους σε άλλες ειδικές επιτροπές, άλλους συναδέλφους σε επιτρόπους διότι ναι μεν η ενέργεια και η οικονομική πολιτική ε, έχει τη θέση της αλλά και άλλοι συνάδελφοι ε, που χειρίζονται θέματα ασύλου, μεταφορών, υποδομών και εκείνοι ε, θέλουν περισσότερο προσωπικό. Το η 5% Ε, πρέπει να, λάβει υπόψη, ε, ε, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν υπάρχουν ανάγκες για περισσότερο προσωπικό. Όμως, εμείς θα παρακολουθούμε τον ΑΣΕΡ και πώς θα λειτουργήσει με τις νέες θέσεις εργασίας και πώς θα αντιμετωπίσει τα καθήκοντά του με το νέο ε, σύστημα τεχνολογίας της πληροφορίας. Και αν σε κανένα δύο χρόνια φανεί ότι δεν έχουν ανταποκριθεί στις ε, αρμοδιότητές τους όπως πρέπει, τότε σε συμφωνία με τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο θα δοθούν περισσότερα κονδύλια. Ε, θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις εκ του σύνεγγης και αυτό σας υπόσχομαι να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε ή έκλεισε η συζήτηση στο σημείο αυτό. Κυρίες και κύριοι, ε, αύριο θα συνεδριάσουμε Τετάρτη ε, στις 9 Οκτωβρίου από τις 9 μέχρι τις 2 και από τις 3 μέχρι τις 11 το βράδυ. Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε και είναι στην διάρκεια